Έκθεση του κυρίου Γκάιερ για περιφερειακή στατηγική για βιομηχανικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι το θέμα. Γιέν Γκάιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά ατμομηχανή για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό φαίνεται ότι και το, από το γεγονός ότι οι χώρες που έχουν ισχυρή βιομηχανική βάση ε, ξεπερνούν τα προβλήματα της κρίσης πιο εύκολα από ό,τι άλλες. Και η Κομισιόν το έχει αναγνωρίσει αυτό. Η στρατηγική για τη βιομηχανία υπάρχει αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο θα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω εγώ είναι η περιφέρεια το περιφερειακό σκέλος της στρατηγικής αυτής γιατί υπάρχουν ορισμένες περιοχές ε, βιομηχανικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ιδιαίτερες ε, ισχύες και ιδιαίτερες αδυναμίες και ιδιαίτερα θετικά σημεία βεβαίως παραδείγματος χάρη στην ε, βιομηχανικές περιοχές όπως αυτή της Λιέγης ή του Ρούρ όπου έχουμε εξόρυξη άνθρακα ή είχαμε εξόρυξη άνθρακα οι συνθήκες ήταν, είναι διαφορετικές από τις άλλες περιοχές επηρεάζεται το περιβάλλον, ιδιαίτερα το έδαφος επηρεάζεται και δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Χρειάζονται δημόσια κονδύλια και μάλιστα πολλά δημόσια κονδύλια. Θέλουμε θα πρέπει οποιαδήποτε παρέμβασή μας να είναι υψηλού επίπεδου. Η όμως τα παραδείγματα που σας έδωσα σχετικά με, την, με τα που έχουν ανθρακοριχεία είναι, δεν είναι οι μόνες περιοχές που έχουν πρόβλημα στην Ευρώπη. Γενικότερα οι βιομηχανικές περιοχές έχουν προβλήματα, προβλήματα σχετικά με ρήπανση και εδάφους και ατμόσφαιρας και από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε. Αυτές αυτή η ιδέα είναι μια γενική ιδέα που με την οποία μπορούμε φαντάζομαι να συμφωνήσουμε όλοι αλλά δυστυχώς ζούμε μια οικονομική κρίση και όσο και να συμφωνούμε με την ιδέα της παρέμβασης μπορεί να μην υπάρχουν οι ε, τα οικονομικά μέσα για να παρέμβουμε όπως τα θέλαμε και γι' αυτό τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Ε, γι' αυτό ζητώ τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκείνους που έχουν πρόβλημα να παρέμβουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου γιατί που με βοήθησαν στην κατάρτιση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. κυρία Κλέβερ. Um, κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση Γκάιερ είναι επίκαιρη, ρεαλιστική, απαραίτητη την επικροτώ λοιπόν και συγχαίρω τον εισηγητή. Η ευρωπαϊκή βιομηχανική πραγματικότητα μας κάνει να δώσουμε μια εγκάρσια εστίαση, μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και επειδή έχουμε το καλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην απαραίτητη αλλαγή μοντέλου ε, να βοηθήσουμε τις βιομηχανικές ζώνες που έπεψαν να, είναι. Γιατί χρειαζόμαστε μια ισχυρή βιομηχανία που θα απευθύνεται προς μελλοντικέ αγορές η έκθεση προσπαθεί να υποφεληθεί και των συνεργειών μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής συνοχής. Πρέπει να προγραμματίσουμε για να έχουμε τα καλύτερα τα αποτελέσματα. Στη χώρα μου όμως δεν, σημαίνει, δυστυχώς, δεν συμβαίνει δυστυχώς αυτό. Αντί να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια, έχουμε κάνει μια ε, δρομολογήση, μια εκπαιδευτική αν θέλετε μεταρρύθμιση ε, που ουσιαστικά θα είναι αναδρομικό και θα διχάσει. Δεν θα προωθήσει ε, ούτε την αριστεία ούτε τις δεξιότητες, κάτι όμως που είναι απολύτως απαραίτητο. Θα πρέπει λοιπόν κυρία Επίτροπη τα περιφερειακά κονδύλια, τα περιφερειακά ταμεία να φροντίσουμε να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, όχι για το διαχωρισμό, τη διαίρεση, αλλά για την ε, επανεκβιομηχάνηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Γιατί με την έκθεσή του ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Η συνθήκη τη Λισαβόνα, τα συστήματα τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και τη οικονομική διακυβέρνηση δεν τα περιλάμβανε λόγω αντίσταση των κρατών μελών, αλλά με την κρίση αναγκαστήκαμε να τα δρομολογήσουμε. Ε, για τον ίδιο λόγο έχουμε μια δειλή αναφορά ε, στη περιφερειακή, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Θα έπρεπε όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη η εστίαση, διότι δημιουργούνται στις περιφέρειες μεγαλύτερη καινοτομία, ανάπτυξη, ε, το δυναμικό και οι βιομηχανικές δεξιότητες ε, είναι, ε, αξιοποιούνται με καλύτερο τρόπο όταν υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους, με τις περιφέρειες. Αυτό το είδαμε και στη χώρα των Βάσκων και ένα από τα σύμβολα που είναι η μεταρρύθμιση, η μεταμόρφωση του Μπιλμπάου αναφέρεται και στην έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να συμπεριληφθούν όταν έχουν μια ταυτότητα οικονομική. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα πρέπει να είναι είναι ένα πρόβλημα, είναι εξαιρετική ευκαιρία, διότι έδειξαν οι τοπικές κοινότητες ότι μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και έτσι από κάτω προς τα πάνω δημιουργείται η Ευρώπη. Σίγουρα η ευημερία ε, και οι πρωτοβουλίε των πολιτών πρέπει να στηριχτούν. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Είναι σύνηθε, αλλά θα δώσω το λόγο σε κάποιον που μίλησε πριν. Κυρία Σάνσε Σμιτ από τη Γαλλία που θέλει ιδιαίτερη βοήθεια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και δεκαετία ο βιομηχανικό τομέα τη Ευρώπη βρίσκεται σε ύφεση. Εστιαζόταν πολύ στι υπηρεσίε και η Ευρώπη λησμόνισε τη βιομηχανία τη και το πληρώνουμε σήμερα το τίμημα η Πεζό, η Continental, η Petro Plus, ο κατάλογο τη πάυση δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ μακροσκελή στη χώρα μου. Απειλούνται οι εργάτε από το κλείσιμο των εργοστασίων. Η μεταγκατάσταση, η ενεργεία του απειλεί και τι θα απαντήσουμε. Η έκθεση δίνει κάποια ίχνη. Δρά και επενδύει η Ευρώπη χάρη στα θετικά ταμεία. 330 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στι περιφέρειε μεταξύ του 2014-2020. Αυτοί θα πρέπει να συνοδεύσουν επίσης τους ανέργους να αναζωογονήσουν τη βιομηχανία, να δώσουν κατάρτιση, να προστηρίξουμε βιώσιμη ανταγωνιστική και ενωτόμα βιομηχανία. Λοιπόν, δημιουργική βιομηχανία και ο πολιτισμό θα πρέπει να οδηγήσει στην αδιάθρωση. ψηφιακή τεχνολογία, υψηλού επίπεδου βιοτεχνία, παραγωγή κινηματογραφική. Είναι πάρα πολλέ δραστηριότητε αυτέ που επιτρέπουν την επαναπροώθηση τη βιομηχανία και να αναζωογονηθεί η επικράτεια. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει τι βιομηχανικέ τη ζώνη η Ευρώπη, θα πρέπει να επενδύσει για το μέλλον του. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μοργάντε, για το λόγο. Ε, πρέπει να τελειώσουμε στις 11. Έχω έναν του ΕΛΚ, ήδη μιλήσατε, έκανα εξαίρεση για την Κέσσανσε Σμιθ, γιατί είναι Γαλλίδα. Διαδικαστικό, ποιο είναι το διαδικαστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, έχω μία ερώτηση. Ποιο κανόνα χρησιμοποιείτε όταν αποφασίζετε ότι είστε μία συζήτηση δεν μπορούν οι ευρωβουλευτές να πάρουν δεύτερη φορά το λόγο. Και σε άλλες περιπτώσεις όμως είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ σημαντική συζήτηση αυτή για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και εμποδίσατε πολλούς ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο μια φορά να δευτερολογήσουν. Αλλά ε, προηγουμένως τους επιτρέψατε να πάρουν το λόγο τρεις ή τέσσερις φορές διαδοχικά. Ποιο κάνω να χρησιμοποιείτε. Απόψε, λέει ο Πρόεδρος. Όλοι μίλησαν μια φορά. Εξαιρετικά δώσα το λόγο στην κυρία Σάνσε Σμποκ που ε, μίλησε ε, εκπρόσωπος της ΕΛΚ αλλά έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Γαλλία του βιομηχανικού τομέα γι' αυτό της έδωσα το λόγο και τον ε, κύριο Μοργκάντη. Άρθρο 149 χρησιμοποιώ. Ο κύριος Μοργκάντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει και σωστά τη σημασία και την αξία τη ευρωπαϊκή βιομηχανία που αντιμετωπίζει σε πολλού τη φαντουργία και χαλιβουργία. Θεωρώ όμω ότι οι λύσει που αναφέρονται δεν λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα τη παρουσία τη βιομηχανική σε μια περιοχή ή την κληρονομιά γνώση και δυναμικού που είναι τυπικό μια περιοχή που αναπτύχθηκε με τον χρόνο. Μιλάμε πάλι για την ευνόηση τη εγκατάσταση πολιτισμικών και δημιουργικών βιομηχανιών που αντικαθιστούν τι παλιέ παραγωγέ. Κατά την άποψή μου δεν είναι αυτή η λύση θα μπορούσαν να είναι κάτι χρήσιμο. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη βιομηχανία που ήδη υπάρχει. Η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τον τομέα της κρουστεφαντουργίας και τη χαλιβουργία διότι υπάρχουν εργοστάσια που επί αιώνες δείξανε ικανότητες που είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αλλού. Στην Τοσκάνη Έχουμε βιομηχανίες προς τη και χαλιβουργία ε, στο Πιομπίνο ε, και αριστεία σε διεθνές επίπεδο στον αφορά την παραγωγή. Και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις βιομηχανίες αυτές και δεν θέλω εκεί η Ευρώπη να θέσει τη λέξη τέρμα πάνω σε αυτές τις βιομηχανίες. Τέλος. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κυρία Γιασνοβέσκα, αν θέλετε γραπτό να υποβάλλετε μια δήλωση. Διότι ήσασταν παρούσα στη συζήτηση. Είναι δικαίωμά σα. Θα αποτελέσει τμήμα τη συζητήσεω. Ο κ. Φεραίρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική που να είναι αξιόπιστη για τις βιομηχανικές ζώνες. Βάσει των υφισταμένων πολιτικών, οι πολιτικές της συνοχής ποτέ δεν είχαν αρκετά χρήματα. Και αυτό επιδεινώνεται με το νεοπολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλε πολιτικές που οδήγησαν στην αποβιομηχανοποίηση, κυρίως στις περιφερειακές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε χρόνιο έλλειμμα και τεράστιο χρέος στις χώρε και επιδεινώθηκε η κατάσταση με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Χρειάζονται σωστέ λύσει. Όχι επιδερμικέ. Χρειαζόμαστε πραγματική βιομηχανική πολιτική για βιώσιμη βιομηχανία, να χρησιμοποιούνται οι πόροι κάθε περιοχή και να ενισχυθούν οι φυστάμενες βιομηχανίε στι διάφορε περιοχέ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπιστούμε τη βιομηχανία των κρατών μελών να απαλλαχθούμε από τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ που δεν βοηθούν καθόλου. Ευχαριστώ. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον αξιότιμο βουλευτή κύριο Γκάιε. Πράγματι αυτή η έκθεση περιέχει πολύ ενδιαφέρουσε πτυχές, είναι και άκρος επίκαιρη. Είναι πολύ σημαντική ιδίω σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής κρίσης και πρέπει ε, να δώσουμε προσοχή ε, στη μάχη ε, που δίνουμε στις παρακμάσουσες βιομηχανικές περιοχές. Επομένως, ε, η χρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών ταμείων είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις μέσω του ERDF στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 7 έως 13 είναι της τάξης των 54,2 δις ευρώ στις 27 κράτη, χώρες μέλη της Ένωσης. Οι περισσότερες επενδύσεις ε, είναι υπέρ της καινοτομίας και πιστεύουμε ότι πολλά από όσα υπόθηκαν στην έκθεση με την καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών συνοχής για τους στόχους του 2020 αντιμετωπίζονται ήδη, όπως και με τις συνέργειες που ελπίζουμε να πετύχουμε, με την ευφυή εξειδίκευση. Βέβαια, χρειάζεται προσπάθεια, ενισχυμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Στο ευρωπαϊκό, στο επίπεδο κρατών μελών, περιφερειακό επίπεδο. Απαιτείται όμω και πραγματική ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε καλύτερες συνέργειες, οδικούς χάρτες. Η έννοια αυτής της ευφυούς εξειδίκευσης, την οποία τα θετικά στην εκθεσή σας, καλή ε, σε στρατηγικές, σε περιφερειακό επίπεδο, προσαρμοσμένες, ε, που θα λαμβάνουν υπόψη ε, το δυναμικό, το αναπτυξιακό και τα θετικά στοιχεία των περιοχών. Πιστεύουμε ότι αυτή η ευφυής εξειδίκευση τρία πράγματα τουλάχιστον μπορεί να κάνει, να στηρίξει την οικονομική μεταρρύθμιση στις ε, αποβιομηχανισμένες περιοχές. Πρώτον, να βελτιώσει τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και αλλαγές να προωθεί σε αναδυόμενες βιομηχανίες, ε, υπηρεσίες προς τις διεθνείς αγορές. Ποτέ την έννοια αυτή, η ευθύης εξειδίκευση μπορεί να θεωρηθεί ε, ως μια ειδική προσέγγιση για την βιομηχανική πολιτική. Δεύτερον, ενίσχυση της μεταφοράς ε, τεχνογνωσίας και γνώσεων με τα ε, ωφέλη που μπορεί να παράσχει σε όλους τους φορείς αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη ε, των κοινωνιών βάσει της ε, ανταλλαγής γνώσεων. Τρίτον, μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός των πολυεπίπεδων πολιτικών έρευνα, τεχνολογία, βιομηχανική πολιτική, πολιτικές βιομηχανικής ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης κτλ. Κινητοποιούνται έτσι φορείς και πόροι σε όλη την περιοχή όταν υπάρχουν κοινοί στόχοι, κοινά οράματα. Τρεις απλά λόγους σας ανάφερα για το τι ε, μπορεί να προσφέρει η ευφύης αυτή εξειδίκευση. Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις ε, για το ΕΤΠΑ. Η υφής εξειδίκευση λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένα μέσο σημαντικό που θα δώσει κίνητρα για την ολοκλήρωση των πολιτικών και θα προωθεί στην οικονομική αλλαγή, τη βιομηχανική ανανέωση που και εσείς ζητείτε στην έκθεση αυτή. Ήδη αρχίσαμε διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους. Συμφώνες τερικών σχέσεων προγράμματα για το 2014 έως 2020. Γίνονται πραγματικά πολύ σοβαρές προσπάθειες ώστε να έχουμε μια εστίαση των προτεραιοτήτων μας σε αυτές τις στρατηγικές για τη μεταμόρφωση αυτών των περιοχών. Ευχαριστώ. Thank you, Thank you, special... Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Γιάννη Σκάιρ για την εξαιρετική έκθεση. Παράγραφος 21. Μήπως θα έπρεπε να προσθέσετε το Σέφιλτ στη δική μου περιφέρεια, γιατί και αυτό χάρη των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και άλλες περιφέρειες του Βασίλειο Βασίλειου, έχει πραγματικά μετασχηματιστεί. Εδώ ολοκληρώνεται στις 8.30 αύριο το πρωί, θα επαναλάβουν οι εργασίες Ολομέλειας. Καληνύχτα σε όλους.